και ε, στη μετάβαση στη δημοκρατία. Ο Πρόεδρος, συνάδελφοι, έχω μία ανακοίνωση που θα σας αναγνώσω στα ε, αγγλικά, ίσως είναι πιο εύκολο για σας. Ο κύριος David Μάρτιν έχει καθυστέρηση την πτήση του και έχουμε την έκθεσή του, η πτήση του έχει καθυστερήσει. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω, αν συμφωνείτε, ε, να συζητήσουμε την έκθεση του κυρίου Μάρτιν, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική για μα. είναι η προσαρμογή του κανονισμού του Κοινοβουλίου στη Συνθήκη τη Λισαβόνα, να τη συζητήσουμε τελευταία απόψε στην ημερήσια διάταξη. Απλώ αλλάζουμε τη σειρά των εκθέσεων. Δεν αλλάζει τίποτα διαφορετικό, ούτε φεύγει. Δεν αλλάζει το περιεχόμενο. Ε, παρακαλώ λοιπόν, επειδή καθυστερεί η πτήση του κυρίου Μάρτιν, να συμφωνήσετε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να είναι παρόν ο εισηγητή μα κατά τη διάρκεια τη ε, συζήτηση τη έκθεσή του. Επειδή είναι επίσημη αλλαγή αυτό της ημερήσιας διάταξης, είμαι υποχρεωμένο να ζητήσω τη συμφωνία του σώματος ε, επ' αυτού. Και ελπίζω να συμφωνήσετε. Thank you very much, colleagues. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ. Yeah. Ναι.